Okay, colleagues. Um, good morning everybody. I suggest that... Καλημέρα. Μου φαίνεται ότι θα αρχίσουμε. Δεν είναι και πολλοί παρόντες, αλλά ο εισηγητής ήρθε και ένας τουλάχιστον από τους κοιόδης. Και αφού είναι 9 και 5 δεν μπορούμε να μην αρχίσουμε. Το πρώτο θέμα είναι το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο της ε, προσφυγές και το δικαίωμα πληροφόρηση κλπ. Η κυρία Ελένη Αντωνέσκου είναι η συγγήτρια. Σήμερα θα εξετάσουμε λέει τις τροπολογίες. Πρόκειται για την τρίτη φάση της εφαρμογής του οδικού χάρτα για τα, δικαστικά ή δικαστικά δικαιώματα Ήδη πέρασαν οι πρώτες δύο φάσεις, γι' αυτό είναι τώρα η τρίτη. Η εισηγήτρια η κυρία Αντωνέσκου υπέβαλε ήδη από το Φεβρουάριο το σχέδιο έκθεσής της και κατατέθηκαν 133 τροπολογίες. Η νομική υπηρεσία δέχτηκε το αίτημα γνωμοδότησης από μας και την εξέταση του θέματος του κατά πόσον είναι συνεπή αυτά που συμβαίνουν στην πράξη με το θέμα των δικαιωμάτων των πολιτών και αν υπάρχει επαρκή και νομικό υπόβαθρο. Με την άδεια της εισηγητρίας λοιπόν, αφού την ακούσουμε να παρουσιάζει τις τροπολογίες, θα δώσω το λόγο στη νομική υπηρεσία. Πριν την ανταλλαγή απόψεων, ναι βλέπω την Εύη η εισηγήτρια, λοιπόν έχει πρώτη το λόγο η κυρία Αντωνέσκου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σωστά είπατε. Πιστεύω και εγώ ότι πρέπει να γίνει η συζήτηση πριν από την ψηφοφορία. Θα θέλαμε η νομική υπηρεσία να μας παρουσιάσει τη γνωμοδότησή της για το άρθρο 12 και το άρθρο 3 της οδηγίας. Αυτά τα δύο άρθρα προβλέπουν κανόνες για τη χρήση των αποδεικτικών στοιχείων που έχουν συλλεχθεί παρανόμως δηλαδή χωρίς τη βοήθεια δικηγόρου. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν και υπέβαλαν τόσο πολλές τροπολογίες. Θα ήθελα να γνωρίζουν ότι θα προσπαθήσω να πετύχω τον καλύτερο δυνατό συμβιβασμό. Για να δούμε τώρα τις τροπολογίες. Για το εύρος άρθρο 2 έχουμε την τροπολογία 85 που λέει ότι για λόγους σαφήνειας πρέπει να λέμε ότι η οδηγία αυτή θα ισχύει όποτε δεν, εφα... δεν δίνονται πλήρη δικαιώματα όποτε μάλλον έχει στερηθεί η ελευθερία του κατηγορημένου. Αυτό το όποτε μπορεί να μας εννοήσει, να μας οδηγήσει να καταλάβουμε ότι οι κανόνες αυτοί ισχύουν μόνο σε περίπτωση σύλληψης. Μετά έχουμε το άρθρο 3 που μιλάει για όλες τις περιπτώσεις που χρειάζεται η βοήθεια δικηγόρου σε περίπτωση σύλληψης. Η κυρία Λάτφορντ κατέθεσε τροπολογία που θέλει να αποσαφινιστεί ότι η οδηγία δεν συμπεριλαμβάνει προ, το, την περίπτωση προανάκρισης της πρώτης προανάκρισης αμέσως μετά τη σύλληψη. Μιλάμε για την προανάκριση που θα καθορίσει αν θα γίνει έρευνα ή όχι. Αυτό το έχουμε συζητήσει στην Επιτροπή μας και κατέθεσα και εγώ μια τροπολογία σχετικώς. Συμφωνώ με την κυρία Λάτφορντ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε στο σκεπτικό και όχι στα άρθρα. Το δικαίωμα σε βοήθεια δικηγόρου το αναφέρει και η τροπολογία 90 δηλαδή. Ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος πρέπει να έχει το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο ενώ το αρχικό κείμενο έλεγε ότι κάθε κράτος μέλος πρέπει απλώς να διασφαλίζει δικηγόρο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν λοιπόν δύο προσεγγίσεις, η δικαιωματική και εκείνη που βασίζεται την ευκαιρία. Ορισμένοι συνάδελφοι ήθελαν να χρησιμοποιηθεί ο, ο όρος επίσημη ανάκριση. Όχι. Σας υπενθυμίζω το εξής. Όταν στη δεύτερη οδηγία για την οδική χάρτα για το δικαίωμα στην πληροφόρηση μιλούσαμε για την ανάγκη χρήσης του όρου επίσημη ανάκριση ή προανάκριση και και λέγω για να καλυφθούν όλες οι περιπτώσεις προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσει ο ύποπτος όταν προανακρίνεται θεωρήσαμε τελικά ότι επειδή είναι διαφορετικοί οι τύποι προανακρίσεων μπορούν να γίνουν δεν χρειάζεται η έκφραση πρέπει ή θα έπρεπε. Για ελάσσονα αδικήματα είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρχει δικηγόρος και πρόσβαση στο τηλέφωνο. Και αυτό στο σκεπτικό και όχι στα άρθρα. Και μόνο όπου δεν υπάρχει περίπτωση δίκης και δεν έχει γίνει σύλληψη. Στο άρθρο 4 για την πρόσβαση σε δικηγόρο και για τη δυνατότητα της παρουσίας του δικηγόρου σε όλες τις ανακρίσεις ή προανακρίσεις. όπου απαιτείται και η παρουσία του υπόπτου Εκεί έχουν κατατεθεί διάφορες τροπολογίες που καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις, τουλάχιστον μία τροπολογία της αναφέρει, συλλογής προκαταρκτικών πληροφοριών ή αποδείξεων. Αλλά δεν τη δέχομαι. Χρειάζεται περισσότερη συζήτηση για αυτό το θέμα. Ελπίζω εδώ να πετύχουμε κάποιο συμβιβασμό. Προτείνω επίσης συμβιβασμό για τη δυνατότητα του δικηγόρου να ελέγχει τις ε, συνθήκες κράτησης και γι' αυτό έχουν κατατεθεί <coughs> πολλές τροπολογίες και νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε μια αποδεκτή λύση να μπορεί ο δικηγόρος δηλαδή να επισκεφθεί τον τόπο κράτησης για να υπάρχει η εγγύηση ότι δεν έγινε η κράτηση χωρίς την άδειά του ή την έγκρισή του. Για τον εμπιστευτικό χαρακτήρα αυτό είναι ιδιαίτερα λεπτό σημείο της οδηγίας και έχουν καταδεχθεί και γι' αυτό πολλές τροπολογίες. Οι συνάδελφοι θέλουν απόλυτο εμπιστευτικό χαρακτήρα στις συζητήσεις μεταξύ πελάτη και δικηγόρου. Άλλοι λένε να υπάρχουν μερικές εξαιρέσεις. Αν υπάρχει σοβαρός λόγος δηλαδή να πιστεύει κανείς ότι ο δικηγόρος συμμετέχει στη διάπραξη εγκλημάτων με συνενοχή, σε συνενοχή με τον ύποπτο ή αν οι δραστηριότητες του μπορεί να βλάψουν τη ζωή κάποιου. moment. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι πρέπει να έχουμε κάποια σοβαρή διαπραγματευτική θέση όταν θα αντιμετωπίσουμε το Συμβούλιο. Έχουν κατατεθεί επίσης πολλές τροπολογίες για τις εξαιρέσεις που προβλέπονται, για τους λόγους που θα τις δικαιολογούσαν με απόφαση βέβαια μιας ανεξάρτητης δικαστικής αρχής και γραπτός. Και εδώ μπορούμε να βρούμε συμβιβάσμα. Όταν κανείς αρνείται το δικαίωμά του σε δικηγόρο, και γι' αυτό έχουν κατατεθεί οι τροπολογίες, πρέπει γραπτός να δηλώνεται αυτό ότι ο ύποπτος δηλαδή αρνείται το δικαίωμά του σε δικηγόρο, γνωρίζοντας όμως τις συνέπειες της δήλωσης αυτής. Η οδηγία θα Ε, τέλεια. Το άρθρο 10. Εδώ θέλω τη γνώμη της νομικής υπηρεσίας. Θα ακούσουμε τα συμπεράσματά της αργότερα. Εδώ το λεπτότερο θέμα είναι η παράγραφος 2. Αλλά υπάρχει το θέμα των ανακρίσεων υπόπτων που τελικά θεωρούνται μετά την ανάκριση ως κατηγορούμενοι. Ό,τι έχουν πει να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια εναντίον τους. Αυτή την παράγραφο ζητούμε να διαγραφεί. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτό αφορά γενικά την ομοθεσία των χωρών μελών και πρέπει να είναι αποκλειστικά εθνικό θέμα θετικό είναι ότι οι συνάδελφοι για το Ευρωπαϊκό Ένταμα Συλλήψεως συμφώνησαν όλοι εκτός από τους Ολλανδούς με αυτή την προσέγγιση. Ε, serviciului Υποβάλαμε στην νομική υπηρεσία ερωτήσεις ως προς δηλώσεις που μπορεί να έχει κάνει ο ύποπτος και τις διάφορες απαλλαγές ή εξαιρέσεις που μπορεί να δεχτεί το σχετικό δικαστήριο, το αρμόδιο δικαστήριο. Υπάρχουν τροπολογίες και προς το σκεπτικό για να υπάρξει μεγαλύτερη συνοχή, αλλά δεν επιμένω σε αυτή, την επιμένω. Υπάρχουν και δύο τροπολογίες που αφορούν τον ορισμό της έννοιας δικηγόρος. Τι είναι δικηγόρος? Και εγώ κατέθεσα σχετικό τροπολογία και υποστηρίζω όλες τις σχετικές τροπολογίες των συναδέλφων σταματάω εδώ για να μπορέσει να μας τα πει και η νομική υπηρεσία. Okay, thank you very much. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ την εισηγήτρια και θα θέλαμε τώρα να ακούσουμε την ε, γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας. Δεν ξέρω ποιος θα μιλήσει εξ της νομικής υπηρεσίας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά την προταθήσα οδηγία σχετικά με την πρόσβαση σε δικηγόρο ε, στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, ετέθησαν δύο ερωτήματα σε σχέση με το, τρία ερωτήματα σε σχέση με τα άρθρα 10 παραγράφος 2 και 13 παραγράφος 3 της πρότασης. Αυτά τα μέτρα είναι αυτά που αφορούν τους λεγόμενους αποκλειστικούς κανόνες, exclusionary rules, ε, οι οποίοι είναι μέτρα που απαγορεύουν την χρήση ε, των, από πλευρά των αρχών ε, των δηλώσεων που έχουν επιτευχθεί από τον υποπτό μετά από παραβίαση των διαδικαστικών δικαιωμάτων. Ε, στην πρόταση της Επιτροπής, ε, τα οι προτινόμενοι κανόνες προσπαθούν να εναρμονίσουν τους εθνικούς ε, κανόνες σχετικά με το παραδεκτό των, των μαρτυριών. Από την άλλη πλευρά, οι προβλέψεις του άρθρου 10 αφορούν την κατάσταση κατά την οποία κάποιος ο οποίος δίνει πληροφορίες στις αρχές γίνεται υποπτός κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και απαγορεύεται η χρήση των δηλώσεών του πριν γίνει ύποπτος. Το άρθρο 13, από την άλλη πλευρά, ασχολείται με την κατάσταση κατά την οποία ένα άτομο το οποίο είναι ήδη ύποπτος πριν ξεκινήσει η ανάκριση δεν έχει δικαίωμα ή του αρνείται η πρόσβαση δικηγόρο ε, και σε, στους κανόνε κανόνες απαγορεύεται η χρήση όλων των δηλώσεων που έχουν γίνει από τον ύποπτο σε αυτή την περίπτωση. Τώρα, να απαντήσω στα ερωτήματα όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, δηλαδή κατά, το πρώτο ερώτημα, κατά, κατά πόσον ε, τα, οι προτινόμενοι κανόνες είναι συμβατοί με τις ε, συνθήκες Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Ε, εκεί θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν και στις συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε και στις συνθήκες λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε στοιχεία τα οποία θα αποβρούσαν να αποτελέσουν πρόσκομα στην έγκριση αυτών των κανόνων. Οι κανόνες ε, στις προτινόμενες οδηγίες ακολουθούν ε, τον στόχο της ε, ε, αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την δικαστική συνεργασία. Επίσης, δεν δημιουργούν οποιαδήποτε, οποιοδήποτε πρόβλημα ή μη ε, συνοχή με τα υπάρχοντα νομικά εργαλεία στο, στην περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σε σχέση με, τον, ε, με τις ποινικές διαδικασίες. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν νομικά εργαλεία στον ποινικό νόμο του Ευρωπαϊκού επίπεδο που να περιορίζουν την δυνατότητα του Ευρωπαίου νομοθέτη να ε, εφαρμόσει αποκλειστικούς νόμους ε, και σε όλες τις περιπτώσεις ε, και όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία και όσον αφορά το ευρωπαϊκό ένταλμα γίνεται τέτοιου είδους συνεργασία. Τώρα όσον αφορά τη νομική βάση της ε, οδηγίας. Θα ήθελα να πω ότι σύμφωνα με την πάγια νομολογία του δικαστηρίου η επιλογή της νομικής βάσης ε, βάση των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται ε, σε, αναφορικά με αντικειμενικά κριτήρια. Αυτοί οι αποκλειστικοί κανόνες ε, όσον αφορά το περιεχόμενό τους είναι κανόνες σχετικά με το παραδεκτό των ε, αποδεικτικών στοιχείων στις ποινικέ διαδικασίες ε, που έχουν σαφέ, σαφή αντίκτυπο στους, στα θεμελιώδη δικαιώματα των υπόπτων. Γι' αυτό λοιπόν εμπίπτουν εις το πεδίο εφαρμογής των δύο διατάξεων του άρθρου 82 που αφορούν δηλαδή τα δικαιώματα των ε, ατόμων στις ποινικέ διαδικασίες και την αμοιβαία αναγνώριση των, ε, και το αμοιβαίο παραδεκτό των μαρτυριών εξειδικεύοντας όσον αφορά τον στόχο του, ε, των κανόνων ε, στην αιτιολογική σκέψη 26 της ε, πρότασης εξηγείται ότι γίνεται σαφής αναφορά στο άρθρο 13 σύμφωνα με τις απαιτήσει που προκύπτουν από την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και επίσης όσον αφορά την δίκαια δίκη υπό το άρθρο 6 του ε, Ευρωπαϊκού ε, Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ε, είναι ανδιαμφισβήτητο ότι οι αποκλειστικοί κανόνες έχουν κάποια επίπτωση στα ε, δικαιώματα των ε, υπόπτων. Αυτό σημαίνει ότι με τους αποκλειστικούς ε, κανόνες δίνεται η δυνατότητα ουσιαστικής εφαρμογής του δικαιώματος που εγγυάται η οδηγία και βεβαίως με τον τρόπο αυτό εφαρμόζεται και το άρθρο 82 κάθετος 2 υποπαράγραφος Β της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ως δικαιονομική βάση. Θα ήθελα υπό το φως των δύο προηγουμένων απαντήσεων να αναφερθώ και στην τρίτη ερώτηση ε, ε, σχετικά με το άρθρο 82.2 υπό παράγραφος α της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει ε, τα μέτρα τα οποία αφορούν το αμοιβαία παραδεκτό των των αποδεκτικών στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών. Ε, αυτό ακολουθεί ακριβώς την ε, διατύπωση των ε, προνοιών της ειδικής λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον χώρο δικαιοσύνης, ασφάλειας και ελευθερίας. Μπορούμε λοιπόν να εξάγουμε ότι τα άρθρα 10 παράγραφος 2, 13, 3 της πρότασης εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 92.2 της ειδικής λειτουργίας και ιδιαίτερα ιδιαίτερα των λιποσημείων α και β. Τέλος, όσον αφορά το κατά πόσο είναι συνεκτική αποκλειστικοί, οι αποκλειστικοί κανόνες ε, με την χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ε, ε, δικαιωμάτων και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η νομική υπηρεσία θεωρεί ότι οι προτινόμενοι κανόνες αντικατοπίζουν ορθώς αυτή την ομολογία. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει ασχοληθεί με τα θέματα αυτά βάσει της υπόθεσης δικαίων διαδικασιών σε μεμονωμένες ποινικέ περιπτώσεις το Δικαστήριο του Στρασβούργου επανειλημμένα θεωρεί ότι το δικαίωμα ε, ενός ε, υπόπτου ή ενός κατηγορούμενου σε, με ποινική διαδικασία ε, να έχει σωστή υπεράσπιση από ένα δικηγόρο είναι ουσιώδες ε, ε, θεμελιώδες μάλλον στοιχείο μιας δίκαιης δίκης. Επίσης ε, έχει καταδειχθεί σε πολλές περιπτώσεις ότι το άρθρο 6 εφαρμόζεται και στην προδικαστική διαδικασία, στις ποινικέ διαδικασίες και ότι θα πρέπει να δοθεί η απαραίτητη νομική αρρωγή στον ύποπτο. Το δικαστήριο υπενθύμησε την σημασία που έχει αυτή η προανακριτική φάση στην προετοιμασία των ποινικών διαδικασιών και έχει αναφέρει ότι το ευάλωτον του κατηγορουμένου ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη. Οποτεδήποτε, ένας, ε, ε, οποτεδήποτε ένα άτομο βρίσκεται σε κατάσταση να θεωρείται ύποπτος δεν θα πρέπει να επιβαρύνεται με την άρνηση της δικαστικής αρρωγής. Όλες αυτές ε, οι αρχές έχουν ε, ε, αντικατοπιστεί στην ομολογία του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι αρχές αυτές οπωσδήποτε δίνουν την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις, τις δυνατότητες αυτές κατά τη διάρκεια της δίκης ο κατηγορούμενος. Τέτοιες οι δηλώσεις οι οποίες θα έχει κάνει επίσης θα, δεν μπορούν να, σε αυτή την περίπτωση να μην ληφθούν υπόψη ως αποδεικτικό υλικό που μπορεί να παρουσιαστεί στο ποινικό δικαστήριο. Ε, αυτά είναι τα κύρια ευρήματα της νομικής υπηρεσίας. Και επομένως, αυτά είχαμε να σας πούμε. Αλλά φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω ε, πρόταση έχετε είτε εσείς προσωπικά είτε άλλα μέλη του, της Επιτροπής σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Έχω έξι που ζήτησαν το λόγο, έξι. Καλά πάμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, πρώτα η Σκιώδης, Ρομέρο Λόπες. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όντως, κάποια από τα προβλήματα τα οποία θέτει ε, αυτό το, αυτή η οδηγία μας τα σημείωσε η κυρία Αντωνέσκου, η συγκήτρια. Ε, και είχαμε και την αποσαφινιστική δήλωση της ε, νομικής υπηρεσίας όσον αφορά τους αποκλειστικούς κανόνες. Τομάδας. Αυτούς τους exclusionary rules που προβλέπονται ε, σε σχέση με την ε, πρόσβαση στον ε, δικηγόρο. Εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια σημεία που πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε συμβιβασμούς. Ήδη έχει δώσει την άποψή της, τη γνώμη της η συγκήτρια, αλλά βεβαίως μπορούμε να συνεχίσουμε την εργασία επί των πλέον αμφιλεγωμένων σημείων, των σημείων αυτών που αποτελούν τριβή Υπάρχουν άλλωστε κάποιες ε, χώρες που ξέρουμε ότι το άρθρο θα είναι ε, πολύ ε, μεγάλο και που δεν περιλαμβάνουν κάτι τέτοιο στην ε, στην ε, νομοθεσία του και εκεί μπορεί να υπάρξουν σημεία τριβής με κάποιες χώρες αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό η γέννηση δικαίου στην προκείμενη περίπτωση να γίνει όσο γίνεται πιο ε, σύντομα, όσο γίνεται πιο γρήγορα και στη διάρκεια των, της προανακριτικής φάσης και στη διάρκεια των ανακρίσεων. Όταν ε, δηλαδή τη στιγμή που ο ύποπτος ε, του δηλώνεται πλέον ότι είναι ύποπτος, γνωρίζει ότι είναι ύποπτος. Θα πρέπει να προχωρήσουμε έτσι ώστε να δούμε ε, τι είναι να μην είναι πλασματικό δίκαιο, ναι, να γίνει πραγματικό δίκαιο να υπάρχει, γιατί έχουμε ας πούμε ε, και την ε, δωρεάν ε, πρόσβαση σε δικηγόρο που δεν λαμβάνεται υπόψη εδώ. Είναι ενδιαφέρουσα και η άποψη της κυρίας Αντωνέσκου όσον αφορά την, το θέμα αυτό. Θα πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να λυθεί και το ζήτημα της δωρεάν ε, πρόσβασης σε δικηγόρο. Τώρα, τώρα. Συμφωνούμε βεβαίως με την θέση της νομικής ε, υπηρεσίας όσον αφορά το ανακριτικό υλικό και ελπίζουμε ότι θα πετύχουμε κάτι καλό και όσον αφορά τις συνθήκες ε, κράτησης. Ξέρετε ότι στις εξαιρετικές περιπτώσεις ε, είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς ε, πότε υπάρχει δυνατότητα κατάρρευσης του απορρίτου ή κατάργηση του απορρίτου μεταξύ ε, του δικηγόρου ε, και του ε, υπόπτου, γιατί καμιά φορά και ο ίδιος ο δικηγόρος μπορεί να είναι υπόπτος και επομένως θα πρέπει να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε και άλλα μέσα έτσι ώστε να επιτύχουμε συγκεκριμένες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε μια παράλληλη διαδικασία. Αλλά βεβαίως αυτές είναι περιπτώσεις ε, περιορισμένες, ε, συγκεκριμένες και θα πρέπει να γίνει μια εις ε, ένας βάθος προβληματισμός γιατί τι θα αναφιβόλω το δικαίωμα υπεράσπισης. Όσον αφορά δε τις καταδικαστικές αποφάσεις ο σκοπός είναι να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό πριν εξάσουμε το ζήτημα των δικαστικών εγγύσεων και είναι απαραίτητο ε, να εξετάσει η Επιτροπή το θέμα αυτό ε, όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικηγόρο. Αλλιώς δεν μπορεί να εξεταστεί παρκώς το θέμα αυτό. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να τηρήσουμε την, ε, το, τις χρονικές προθέσεις, το χρόνο μας. Εγώ ίδια θα επιδείξω αυτοπιθαρχία. Αλλά παρακαλώ και εσείς να τηρείτε τα χρονικά όρια. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Μούλτερ εκ μέρους των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλάω εξ ονόματος της Σάρας Λούτφορντ. Έχω μπροστά μου το κείμενό της γιατί δεν μπορεί να έρθει η ίδια. Δεν σημαίνει όμως ότι τα πιστεύω κι εγώ όλα αυτά. Λέει, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η εγγύηση του δικαιώματος ε, αρρωγής από δικηγόρο. Ελπίζω να συμφωνήσει η Επιτροπή μας ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Επίσης πρέπει η αστυνομία να μην έχει το δικαίωμα να ανακρίνει κάποιον υποπτώ μετά από κάποιο σημείο χωρίς την αρρωγή δικηγόρου. Νομίζω ότι η, όταν είμαστε βέβαιοι ότι γίνεται ότι ετοιμάζεται συλλογή αποδείξεων για προσαγωγή σε δίκη πρέπει οπωσδήποτε να έρχεται δικηγόρος. Καλό θα ήταν να δεσμευτούν τα κράτη-μέλη και να μην επαναλαμβάνουμε απλώς αυτά που λέει η σχετική σύμβαση για τον εμπιστευτικό χαρακτήρα. Φαντάζομαι ότι όλα τα κράτη συμφωνούν. Αλλά παρά τη γενική αυτή συμφωνία, ως γνωστόν ο διάβολος βρίσκεται ελοχεύει στις λεπτομέρειες και υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο δικηγόρος σαφώς δίνει σημεία ότι είναι συνένοχος με τον ύποπτο. Όσο για την αποτελεσματικότητα της οδηγίας και την απαγόρευση χρήσης των αποδεικτικών στοιχείων από την προανάκριση σε δικαστήριο, νομίζω ότι το δικαστήριο είναι το αρμοδιότερο να αποφασίσει. Ξέρω από την νομική μας υπηρεσία ότι αν θέλουμε μπορούμε να νομοθετήσουμε σχετικώς αλλά χρειάζεται περισσότερη συζήτηση χωρίς αυτό να προδικάζει ή να υποβιβάζει το δικαίωμα κάθε δικαστηρίου να καθορίζει τα πράγματα. Αλλά βέβαια δεν μπορεί να αποκλειστεί καρά σε πολύ συγκεκριμένες και ελάχιστες περιπτώσεις το δικαίωμα τηλεφωνήματος σε δικηγόρο και η αστυνομία πρέπει να μπορέσει και αυτή να μας πει πριν ασχίσει να ισχύει η οδηγία τι θέλει να ισχύει. Αυτά είχε να πει η κυρία Λούτφορντ και επειδή μόνο εμπνεύματι είναι παρούσα, πάει έκανα εγώ την παρουσίαση. Έχω όμως και εγώ να προσθέσω κάτι. Έχω καταθέσει τροπολογίες που λένε κυρίως ότι δεν πρέπει να υπερβάλλουμε στην οδηγία για κάθε πλημέλημα να ζητιέται συστηματικά δικηγόρος, να υπάρχουν όρια. Ευχαριστούμε. Πολύ καλά εκπροσώπησες τη Σάρα. Από τους Βαγευράσινους ο Αλμπρέχτ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Αντωνέσκου για την έκθεση της και το συντονισμό των προσπαθειών για την εξέβρεση συμβιβασμού. Επίσης νομίζω καλό ήταν που ζητήσαμε γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου. Έχω τρία σχόλια. Πρώτον, συμφωνώ απόλυτα ότι δεν είναι σωστή η έννοια της επίσημης προανάκρισης. Καλύτερα να μείνουν τα πράγματα όσοι είχαν γιατί αλλιώς μπορεί να γίνουν να σημειωθούν παρερμηνίες. Νομίζω πίσω ότι μας το ξεκαθάρισε η νομική υπηρεσία ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επίσης καθόρισε κριτήρια μιας δίκαιης δίκης. Και αυτά που λέει το άρθρο 6 περιορίζονται στις πρώτες φάσεις μιας ανάκρισης. Δεν θα ήταν σωστό να περιορίσουμε το εύρος του όλου πράγματος, γιατί τότε θα βγαίναμε εκτός θέματος. Για τη συλλογή των αποδείξεων και το θέμα της εμπιστευτικότητας, καλά τα λέει, ιδίως στο 12, όπου όμως θα προτιμούσα να τηρηθεί η παλιά ορολογία, η αρχική ορολογία. για τον εμπιστευτικό χαρακτήρα κάθε. Νομίζω ότι δεν πρέπει να νερώσουμε, να αποδυναμώσουμε την έννοια αυτή γιατί είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει αυστηρή εμπιστευτικότητα και να μην αφήσουμε ανοίγματα και υπερβολικά πολλές εξαιρέσεις. Τέλος, για αυτά που, λένε, που λέει το άρθρο 13.3, συμφωνώ με την νομική υπηρεσία. Υπάρχουν σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν τις ρήτρε αυτές για να υπάρχει μια συνέπεια στο δικαίωμα, στα δικαιώματα των υπόπτων και για να εφαρμόζεται και η ισχύουσα νομολογία. Παρακαλώ λοιπόν γενικά να παραμείνουμε στην ισχύουσα ορολογία, ιδιαίτερα σε αυτή την παράγραφο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κύρκοπ. Ευχαριστώ, πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για το έργο της και θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι πολύ με, ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Υπάρχουν κάποια θέματα και χαίρομαι που η νομική υπηρεσία τα εξέτασε. Και μιλώντας σαν ε, δικηγόρος θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που τονίζουμε ιδιαίτερως την ανάγκη να εξασφαλίσετε πρόσβαση όχι μόνο σε δικηγόρο, αλλά να μπορεί να κοινοποιείται η σύλληψη από τον ε, συλλευθέντα προς κάποιον πρόσωπο της επιλογής του, για παράδειγμα τον εργοδότη του, ούτως ώστε να γνωστοποιείται το γεγονός πριν ακόμα συναντηθεί με τον δικηγόρο. Θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως δικαίωμα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ιδιαίτερος σημαντικό. Επίσης το δικαίωμα βεβαίω, να επικοινωνήσει κανείς με τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές αν κανείς δεν διαμένει στη χώρα καταγωγής τους. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι περιορισμένο το έπρο των παρεκκλήσεων. Η πρόσβαση θα πρέπει να αρνείται μόνο στην περίπτωση όπου υπάρχει ζήτημα δικονομικών εγγύσεων ή αποδεικνύεται αυτή η αναγκαιότητα γιατί θεωρώ ότι είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα η προσφυγή σε δικηγόρο. Η βελτίωση είναι επίση το δικαίωμα να μιλάει κανεί με το δικαιώμα στο τηλέφωνο. Εμεί ασκήσαμε σχετικά πιέσει, γιατί πάντοτε δεν είναι δυνατόν να έχει κανεί άμεση επαφή με το δικηγόρο και αυτό χρησιμοποιείται σαν άλλο για να στερήσει κανεί τον κατηγορούμενο από τα δικαίωμα επαφή. Και αυτό είναι απολύτω απαράδεκτο στι σύγχρονε κοινωνίε με την πρόοδο των τηλεπικοινωνιών. Ε, για παράδειγμα τη διάρκεια της νύχτας ή μια, ε, στην Ήπεθρο όπου είναι μεγάλε οι αποστάσει. Τουλάχιστον μπορεί να γίνει η επικοινωνία εξασφαλιστή με το τηλέφωνο. Θεωρώ ότι αυτό συνιστά μεγάλη βελτίωση. Νομίζω ότι η χρονική περίοδο, όσο το αναλάβει δράση ο δικηγόρο και ε, η παροχή νομική συμβουλή. Νομίζω ότι είναι σημαντικό όσον αφορά τη συγκέντρωση αποδεικτικών ε, στοιχείων. Ε, Εμεί δεν θέλουμε να γίνει οτιδήποτε παρεμποδίζει την ε, διεξαγωγή της ε, ερευνητικής διαδικασίας. αλλά υπάρχει η ανάγκη επαρκούς συγκέντρωση αποδεκτικών στοιχείων και νομίζω ότι ακριβώς αυτό είναι το σημείο της ισορροπίας. Ε, κύριε Πρόεδρε, σε γενικές γραμμές θεωρούμε ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία και βεβαίως θα συνεχίσουμε να δίδουμε την πλήρη μας υποστήριξη. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος, η κυρία Ζίπελ, ευχαριστώ πολύ και εγώ θα προσπαθήσω να περιστώ σε δύο-τρία σημεία και θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο της και φαντάζομαι ότι θα πρέπει να κάνει πολλές συζητήσεις με όλους τους συγκητές τους ώστε να έχουμε μια ισχυρή ε, διαπραγματευτική θέση. Τα τρία σημεία έχουν ως εξή. Καταρχήν το δικαίωμα σε δικηγόρο, ε, πρόσβαση σε δικηγόρο. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορούμε να το περιορίσουμε, έστω και αν πρόκειται για ελάσσον ε, αδίκημα, ε, για το οποίο κανείς δεν έχει, για μια παράβαση για παράδειγμα δική. και θεωρείται καμιά φορά ότι θεωρείται η προσφυγή σε δικηγόρο ότι βαραίνει το αδίκημα, αλλά αυτό δεν ισχύει, δεν θα πρέπει να είναι έτσι. Τώρα, ποια είναι, πώς ε, εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε δικηγόρο. Εγώ προσωπικά δεν έχω δικηγόρο. Ε, δεν μπορώ τηλεφωνικά να απευθυνθώ σε δικηγόρο που είναι ένας εντελώς ξένος σε μένα άνθρωπος. Θεωρώ ότι θα πρέπει να μπορεί ο ύποπτο να επιλέγει προσωπικά τον τρόπο επαφής με τον δικηγόρο του. Τώρα, όσον, όταν, όσον αφορά την παρέτηση από το δικαίωμα προσφυγή σε δικηγόρο, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αναθεώρησης αυτού του, δικαιωμα, του δικαιώματος. Θα πρέπει αυτό να είναι αναστρέψιμο και εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να περιορίζεται η εμπιστευτικότητα γιατί μόνο η εμπιστευτικότητα εξασφαλίζει μια δίκαιη δίκη. Και αυτό ισχύει και για το ζήτημα ελέγχου των συνθηκών κράτησης. Και εγώ ίδια θα ήθελα να παρατηρήσω εδώ ότι πιστεύω το ζήτημα των συνθηκών κράτησης αλλά και επίσης της ε, διάρκειας της ε, προκράτησης θα πρέπει να είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ρυθμιστεί μεταξύ των χωρών μελών. Και ένα τελευταίο σημείο είναι η συνεκτικότητα των διαφόρων μέτρων στον οδικό χάρτη. κυρία Αντωνέσκο αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα και νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικότερα το κείμενο για να μην καταλήξουμε σε εντελώ διαφορετικέ μεταξύ διατυπώσεις των διαφόρων μέτρων. Και θα ήθελα να σε επισημάνω το εξή ε, κάπως με ενόχλησε το γεγονός ότι τα μέτρα αυτά στη γερμανική μετάφραση ε, αναφέρονται ως εξής το δικαίωμα σε, δικα... σε ε, αρρωγή. Εμείς πάντοτε στα γερμανικά λέγαμε ε, το δικαίωμα προσφυγής σε δικηγόρο, όχι σε δικαστική αρρωγή. Δεν θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να εισάγονται εντελώς νέες ε, έννοιες ο κύριος Φώσο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω δύο σύντομες ε, παρατηρήσεις σχέση με τόσο είπε η κυρία Ζίπελ. Εάν ψάχνετε δικηγόρους, ο Τιμόθε και εγώ ίδιος μπορούμε να σας βοηθήσουμε. Τώρα, όσον αφορά το τίτλο στα γερμανικά, θα έλεγα ότι θα πρέπει να εξασφαλίσετε πρόσβαση στην ναι. παράσταση του δικηγόρου ή στο δικηγόρο κλπ. Και ήδη κατ' επανάληψη είπα ότι γενικώ με ικανοποιεί το κείμενο της ε, Κομισιόν. Και όσον αφορά το σχέδιο έκθεσης της Έλενα, ε, επίσης είμαι ικανοποιημένος γιατί ε, είναι πολύ δύσκολο σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα να συνδυάσει κανείς όλα τα στοιχεία. Ιδιαίτερα επειδή οι νομικές παραδόσεις αλλά και και πρόκειται για μια παρέμβαση στο δικονομικό δίκαιο των χωρών. Και όταν ε, ε, και η συνοχή της ε, σύλληψης όταν ο ύποπτος κάνει μέσα στη σπουδή του κάποιες πρόχειρες επιπόλες δηλώσεις θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να διορθωθεί αυτό και να ενταχθεί στην κανονική διαδικασία. Ένα άλλο σημείο το οποίο θα έπρεπε να σκεφτούμε η εξέταση των συνθήκων κράτησης, ε, προφυλάκησης. Ε, νομίζω ότι αυτός ο έλεγχος των συνθήκων κράτησης δεν μπορεί παρά να αυξήσει την ασφάλεια δικαίου. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποια ένσταση εδώ. Και υπάρχουν πάρα πολλές ε, τροπολογίες που αναφέρονται ακριβώς στην ανάγκη διατήρησης του ελέγχου των συνθήκων κράτησης. Δεύτερο σημείο είναι το άρθρο 10 παράγραφος 2 και άρθρο 13 παράγραφος 3. Νομίζω ότι το στοιχείο αυτό θα πρέπει να διαγραφεί από την οδηγία. Ενδεχομένω να είναι σωστά τα όσα είπε η νομική υπηρεσία. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα ανταπιχείρημα εδώ. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχει ρύθμιση εδώ αναγκαίο και θεωρώ ότι δεν υπάρχει απόλυτη ανάγκη να ρυθμιστεί κάθε λεπτομέρεια γιατί ακριβώς παρεμβαίνει στις παραδόσεις των διαφόρων χωρών και είναι ζήτημα, αντίθετο ζήτημα εδώ της αξιοποίησης των αποδεικτικών στοιχείων. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αφήσει κανείς κάποια διακριτική ευχαίρεια στις χώρες μέλη, εν σχέση με τη διαδικασία που επιθυμούν να ακολουθήσουν. Τώρα, όσον αφορά την εμπιστευτικότητα, θα έλεγα ότι και στη θέση με τον δικηγόρο υπάρχει, υπάρχουν περιθώρια να γίνουν καταχρήσεις δηλαδή να υπάρχουν δικηγόροι οι οποίοι ήδη εμπλέκονται σε κάποιες ε, ποινικέ διαδικασίες ή βαρύνονται με κάποιες κατηγορίες. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να υπάρξει ένας επακριβής ορισμός με κάποια δυνατότητα εξαιρέσεων, ούτως ώστε να αποφεύγονται αυτές οι δυνατότητες κατάχρησης εκ μέρους των δικηγόρων. Τώρα, Όσον αφορά την τροπολογία 126 της κυρίας Ζίπελ και ο κύριος Άλμπρεχτ ε, αναφέρθηκε εδώ, την εξασφάλιση μιας δίκαιης διαδικασίας και την αποφυγή των βασανιστήριων και της απάνθρωπης μεταχείρισης. Μου φαίνεται εντυπωσιακό ότι θα μπορούσαν ε, τα βασανιστήρια ή η απάνθρωπη μεταχείριση των κρατουμένων να είναι κομμάτι της καθημερινότητας της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν, μπορώ, δεν το ζήτημα των ε, παραδόσεων της CIA. Θα ήθελα να καλέσω την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μας παρουσιάσουν εν συντομία τις παρατηρήσεις τους και να τις περιορίσουν στο απολύτως αναγκαίο. Γιατί θέλω να τηρήσω το σημερινό χρονοδιάγραμμα και να δώσω και το λόγο στην εισηγήτρια. Καταρχήν από την Επιτροπή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Αντωνέσκου, την εισηγήτρια για τις παρατηρήσεις τις οποίες καλωσορίζουμε κυρίως ε, όσον αφορά την εμπιστευτικότητα των ε, ε, ανακρίσεων. Επίσης, και υπό το φως συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση η Κομισιόν πέρα από τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί χαιρετίζει μια γενική τάση του Κοινοβουλίου ε, που εκφράζουν θέληση αφενός να δεχτούν την οδηγία και δεύτερον ε, να προχωρήσουν σε αυτόν τον δρόμο που δείχνει η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έτσι ώστε να δείξουμε ε, τον δρόμο όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικότερα και το δικαίωμα στην εισπεράσπιση ειδικότερα. Όσον αφορά τις κυρώσεις, άρθρο 13 η Κομισιόν συμμερίζεται την άποψη της ομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου με μία επιφύλαξη. Δηλαδή ότι η Κομισιόν θεωρεί ότι στρίκτο σένσου δεν ε, ε, ενέχονται εδώ ε, οι κανόνες του παραδεκτού των μαρτυριών ή των αποδεικτικών στοιχείων, αλλά μία γενικότερη αποδοχή των ε, ε, στοιχείων και ότι ο Εθνικός Δικαστής θα έχει τη διακριτική ευχέρεια ε, να συμπεριλάβει τα στοιχεία αυτά ή να τα αποκλείσει κατά την περίπτωση κατά την οποία τα στοιχεία αυτά ενδεχομένως αλλοιώσουν το δικαίωμα που έχει ο κατηγορούμενος για δίκαιη αντιμετώπιση. Εν πάση περιπτώσει ε, ε, κανένα δίκαιο δεν είναι πραγματικό εάν ε, δεν έχει τις εξαιρέσεις του σε περίπτωση παραβίασής του και επομένως εμείς θεωρούμε ότι αυτή ε, η διάταξη θα πρέπει να διατηρηθεί στο τελικό κείμενο και ε, ε, με τον τρόπο αυτό ο εθνικός δικαστή ή υπό τον έλεγχο βεβαίως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να έχει την δυνατότητα να αποφανθεί εάν και κατά πόσον έχει υπάρξει παραβίαση του δικαιώματος. Ευχαριστώ πολύ. Σόλκοφ από τη Δανική Προεδρία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να πω εξ ονόματος της Προεδρίας ε, ότι βρίσκω τη συζήτηση αυτή, καθώς επίσης και τις τροπολογίες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες το Κοινοβούλιο ε, κατανόησε αμέσως ότι πρέπει να βρεθεί ε, μια σωστή ισορροπία και αυτό αποτελεί καλή βάση για, για μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Ε, δεν έχω εντολή αυτή τη στιγμή να κάνω οποιαδήποτε σχόλιο όσον αφορά τις προτάσεις του Κοινοβουλίου, διότι το Συμβούλιο ακόμα βρίσκεται σε διαδικασία συζήτηση έτσι ώστε να καθορίσει τη δικιά του διαπραγματευτική διαπραγματευτική ε, γραμμή και διαδικασία. Ούτε αυτό είναι εύκολο βέβαια γιατί στα κράτη-μέλη οι εθνικοί νόμοι διαφέρουν και μερικές φορές διαφέρουν ουσιοδός όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Επομένως ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει την εργασία. Πάντως ε, η Ιδανική Προεδρία θεωρεί ότι ε, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις στα πλαίσια της Δανικής Προεδρίας ακόμα. Γι' αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον ε, θα παρακολουθήσω την έκβαση των διαπραγματεύσεων και στο Κοινοβούλιο, γιατί πρόκειται ένα πάρα πολύ, για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, σημαντικό ζήτημα. Ε, δεν νομίζω ότι έχω να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Επομένως, ε, επαναρχόμαστε στην κυρία Αντωνέσκου, την εισηγήτρια, αν θέλει να κάνει τις τελικές της παρατηρήσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις παρεμβάσεις τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και την νομική υπηρεσία ε, γιατί ε, μας έδωσε μια κατευθυντήρια γραμμή για τις για τις ε, μελλοντικές ε, ε, συζητήσεις. Είναι πολύ σημαντικά τα σημεία τα οποία αφορούν το παραδεκτό και την χρήση των μαρτυριών και των αποδεικτικών στοιχείων. Νομίζω εδώ θα πρέπει να βρούμε κάποια, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε συμβασμό όσον αφορά τα ένδικα μέσα. Πρέπει να εδώ και από κοντά όλα τα ζητήματα τα οποία έθιξαν. Το γεγονός ότι δεν ανέφερα ε, την ε, ε, δωρεάν νομική αρρωγή δεν σημαίνει ότι δεν με ενδιαφέρε το θέμα. Θα ήθελα να πω λοιπόν στην κυρία Ρομίρο Λόπες ότι μαζί με τον κύριο Σάιμον Μπουζουτήλε ζητήσαμε από την Επιτροπή να προχωρήσει η τροποποίηση του κειμένου ε, που θα αφορά ακριβώς ε, την ε, ενδυνάμωση του δικαιώματος της δωρεάν παροχής νομικής αρρωγής. Θα ήθελα να πω στους συναδέλφους μου ότι είναι προφανές ότι χρειαζόμαστε σαφή θέση έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε. Δεν είναι δυνατόν απλώς να έχουμε απλώς ε, τη θέση του Συμβουλίου, θα πρέπει να έχουμε και μια δικιά μας θέση για τις διαπραγματεύσεις. Επομένως, ε, θα ήθελα να ζητήσω από όλους ε, συνεργασία. Να σας ζητήσω λοιπόν να με βοηθήσετε έτσι ώστε να φτάσουμε στην καλύτερη δυνατή διαπραγματευτική θέση όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Η κυρία Σίπελ έχει δίκιο πρέπει να ορίσουμε σε συνεργασίες, σε συναντήσεις με τους συναδέλφους, με τους κοιόδης συγητής για να μπορούμε να βρούμε αυτά τα ισχυρά σημεία και ενδεχομένως θα πρέπει να ε, μεταθέσουμε την ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία λέει η Πρόεδρος. Επομένως ολοκληρώσαμε την εξέταση αυτού του σημείου της ημερησία διατάξεως και επομένως μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Βλέπω ότι ο κύριος Μπουζουτήλ δεν είναι εδώ. Hmm. Προτείνω πάντως να ξεκινήσουμε ήδη. Okay. Um, point 12 the agenda. Σημείο 12 στη μέση διάταξη. Απόφαση του Συμβουλίου για τη συμπλήρωση του κώδικα συνόρου των, ε, του Σέγγεν όσον αφορά την επιτήρηση των εξωτερικών θαλασσίων συνόρων στα πλαίσια της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από την Frontex. Το 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να ε, αντιταχθεί στην ε, απόφαση αυτή και θα καλέσουμε τώρα την νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μας παρουσιάσει τα συμπεράσματα του Γενικού Εισαγγελέα στην υπόθεση και μετά θα ακούσουμε και την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του εισηγητού και όποιου άλλου θέλει το λόγο. Ε, η κυρία Ντίν, από ό,τι κατάλαβα, θα είναι εδώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εσείς ζητήσατε τη γνωμοδότηση αυτή. με θέμα την επιτήρηση των θαλάσσιων εξωτερικών συνόρων στα πλαίσια τη ψυχιακή συνεργασία που συντονίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση τη Επιχειρηματική Συνεργασία Εξωτερικά Συνόρων των Κρατών Μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Frontex. Και η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν είχε τότε μαζευτεί. Στις 17 Απριλίου 12 ο Γενικός Εισαγγελεύς γνωμοδότησε και υποστήριξε τη θέση του Κοινοβουλίου. Πρώτα πρώτα θα ήθελα να πω ότι η γνωμοδότηση αυτή δεν είναι δεσμευτική για το δικαστήριο και δεν είναι αναγκασμένο να την ε, δεχτεί. Αλλά αποτελεί μία πλήρη ανάλυση των στοιχείων παρόλα αυτά. Στη γνωμοδότηση του ο Γενικός Ισαγγελεύς έθιξε δύο θέματα. Κατά πόσο είναι αποδεκτό αυτό που έγινε η απόφαση του Συμβουλίου, δηλαδή κώδικας για τα σύνορα και ποια είναι τα ουσιώδη και μη ουσιώδη στοιχεία. Πρώτον για το αποδεκτό, παραδεκτό. Το Συμβούλιο είπε ότι επειδή το Κοινοβούλιο είχε λέει υπερβεί τις δικαιοδοσίες του, δεν έχει τώρα το δικαίωμα να προσφύγει για τον ίδιο λόγο. Ο Γενικός Εισαγγελεύς το απέρριψε αυτό, επειδή το Κοινοβούλιο δεν υποχρεωμένο να αντιταχθεί σε μία πράξη ακόμη και αν έχει δικαίωμα να ασκήσει αρνηση κυρία, μπορεί η θέση του να εξαρτάται από πολιτικές, από πολιτικά κριτήρια και η άσκηση του βέτο δεν είναι τίποτε το υποχρεωτικό. Άρα η άσκηση της κυρίας και το δικαίωμα να αμφισβητήσει κάποια νομική πράξη είναι δύο ανεξάρτητα πράγματα. Αυτό κατά τον Γενικό Εισαγγελέα φάνηκε και από τη διαδικασία. Για να ασκηθεί το βέτο του Κοινοβουλίου στην κανονιστική διαδικασία πρέπει να υπάρχει πλειοψηφία των μελών, όχι των παρόντων, αλλά των ε, μελών του Κοινοβουλίου. Ενώ για να γίνει προσφυγή στο δικαστήριο δεν χρειάζεται καν ψήφος της, πλειο... της Ολομελίας. Άρα η δυνατότητα τα άσκησης ε, αγωγής για την κατάργηση κάποιας νομικής πράξης είναι δυνατή. Στην περίπτωσή μας προβλεπόταν η έγκριση από την Κομισιόν πρόσθετων μέτρων, α όχι όχι, πρόσθετων μέτρων για την επιτήρηση σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία το Κοινοβούλιο έλεγε ότι η απόφαση περιελάμβανε στοιχεία ουσιώδη και άρα ότι αφορούσαν τον νομοθέτη. Ο Γενικός Εισαγγελεύς εξέτασε γενικά την, ε, τα πράγματα και είπε ότι τα όρια πρέπει να τεθούν από το χαρακτήρα της αμφισβήτησης και είπε ότι εδώ ο τομέας πολιτικής, δηλαδή ε, επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων, αφορά και τα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τελείως τεχνικά θέματα όπως την πολιτική γεωργίας, όπου η Κομισιόν γενικά έχει τις περισσότερες αρμοδιότητες και γι' αυτό η νομολογία πρέπει να θεωρείται με φρόνηση. Ε, το κατά πόσο είναι ουσιώδης χαρακτήρας δεν είναι κάτι το μηχανιστικό με βάση απλώς την ομολογία αλλά πρέπει να προκύπτει από μία αξιολόγηση όλων των παραγόντων. Το στόχο της νομοθεσίας κλπ. Άρα πιστεύει ότι η απόφαση αποτελεί νέα ουσιώδη στοιχεία τα οποία συμπεριλαμβάνουν την πρόσβαση σε κάποιο πλοίο, την κατάσχεσή του, την παράδοσή του σε αρχές τρίτης χώρας και κατά αυτόν οι ρήτρε ως προς το που πρέπει να γίνει η αποβίβαση αποτελούν επίσης νέα ουσιώδη στοιχεία για την επιτήρηση των θαλασσίων εξωτερικών συνόρων και δίνει τους εξής λόγους τα μέτρα αυτά απαιτούν δύσκολες αποφάσεις που σχετίζονται με την προσωπική ελευθερία των ενδιαφερομένων, τη δυνατότητά τους να τύχουν διεθνούς προστασίας και μπορούν να επηρεάσουν και τη σχέση με τρίτες χώρες. Εκτός αυτού η δυνατότητα εφαρμογής τέτοιων μέτρων στην ανοιχτή θάλασσα είναι κάτι ανεξάρτητο από τον κώδικα των συνόρων του Χσέγγιν. Δύο άλλα στοιχεία δείχνουν ότι είναι ουσιώδη τα μέτρα αυτά πρώτον θέτουν θέματα ιδιαίτερα λεπτά και αμφιλεγόμενα όπως την εφαρμοσιμότητα ή μη της ε, επαναπροώθησης όσων θα αποβιβαστούν και δεύτερον τον καθορισμό συγκρίσιμων στοιχείων σε σχέση με την ομολογία. Ο Γενικός Ισογγελέα επίση δέχτηκε το επιχείρημα του Κοινοβουλίου ότι η απόφαση αυτή αφορά τη συνεργασία στα πλαίσια του πρόντεξ και ότι όλα αυτά ξεπερνούν τις δικαιοδοσίες που χορηγούνται στον κώδικα του Σέγγεν. Ιδιαίτερα αυτά που προβλέπει η δεύτερη προσθήκη για τις αποβιβάσεις που δεν προκύπτουν από το Σέγγεν αλλά από το συγκεκριμένο επιχειρησιακό πλαίσιο και ότι δεν απαιτείται τροποποίηση των κανόνων του Σέγγεν. Ο Γενικός Εισαγγελέφης επομένως προτείνει την ακύρωση της απόφασης αλλά τη διατήρησή της μέχρι την έγκριση σχετικού νομοθετήματος. Εάν το δικαστήριο ακολουθεί στην άποψη του Γενικού Εισαγγελέα, τότε πρέπει να προταθεί αντικατάσταση της απόφασης του Συμβουλίου με άλλη πράξη που θα εγκριθεί με την κανονική, με τη συνήθη διαδικασία. Και μπορούμε να ελπίζουμε ότι η απόφαση του δικαστηρίου θα αποτελεί μια χρήσιμη καθοδήγηση για όλα τα όργανα ως προς τον διαχωρισμό ουσιωδών και μη ουσιοδών στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 290. Αυτά είναι τα κύρια στοιχεία της γνωμοδότησης του Ισαγγελέα και είναι διαθέσιμη, είμαι διαθέσιμη για τυχόν απορίες και παρεξηγήσεις. Ωραία λοιπόν, θα ακούσουμε την Επιτροπή, εν συντομία την κυρία Έμα Μπράουν, εφόσον το επιθυμείτε, όχι. Τότε θα περάσουμε στον κύριο Κάσμαν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε Μάγκη για την εξαίρετη ανάλυση σου. Χαίρομαι πάρα πολύ που ε, τονίζει τη θέση την οποία εγώ ε, παρουσίασα, έστω και αν η Επιτροπή δεν την αποδέχτηκε. Ιδιαίτερος όσον αφορά το αποδεκτό στην παράγραφο 3, όπου ο Γενικός Εισαγγελέας δηλώνει ότι η διαδικασία μπορεί να υπαχθεί σε κάποιους προβληματισμούς πολιτικής ε, φύσεως. Και αυτό ακριβώς επεσήμενα το πλαίσιο της απόφασης λέει ότι οι χώρες μέλη θα πρέπει να ε, μείνουν πιστές στις εθνικές αρχές όσον αφορά το ναυτικό δίκαιο. Και ε, υπήρξε ενδίδραση της Μάλτας και της Ιταλίας, γιατί οι κανόνες λένε ότι η κανονικοί ότι οι μετανάστες οι οποίοι διασώζονται από τις υπηρεσίες της ε, Frontex υπάγονται στην ε, νομοθεσία της ε, χώρας υποδοχής. Και όλοι όσοι σώζονται άρα λοιπόν από τη Frontex της Μάλτα θα πρέπει να εμφανιστούν στις αρχές της Μάλτας. Θεωρώ ότι η Επιτροπή έχει υπερβεί τις αρμοδιότητές της και η βασική μου, το βασικό μου επιχείρημα ε, δεν είναι δυνατόν οι νομικές διαμάχες να γίνονται εις βάρος των ανυπεράσπιστων ε, μεταναστών που πνίγονται στη θάλασσα. Εν πάση περιπτώσει, η δική μου σύσταση δεν ε, υιοθετήθηκε και πήγε στην Ολομέλεια. Όπως ακούμε ότι δεν πέτυχε την ειδική πλειοψηφία. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Μπουσατήλ, ο ξότιμος συνάδελφος, επανήλθε στην Επιτροπή με το αίτημα να αποφανθούν η νομική υπηρεσία κατά πόσο θα μπορούσε ο κανονισμός να απορριφθεί για με το επιχείρημα ότι η Κομισιόν υπερεύει τις αρμοδιότητές της. Αλλά επίσης συμφωνήθηκε ότι η απόφαση στην οποία συμφώνησε η Επιτροπή δεν θα έπρεπε να ανασταλεί. Και χαίρομαι που ο κύριος Μπουσατήλ ε, συμφώνησε στην ε, αναθεώρηση της, ε, για την αναθεώρηση της Frontex και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να τον ευχαριστήσω όχι όσον αφορά το σύνολο. Τώρα, ε, χαιρετίζουμε τη γνωμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα και επίσης ε, θα ήθελα να πω ότι είμαι ιδιαίτερο σύμφωνος με το γεγονός ότι η σύσταση του Γενικού Εισαγγελέα βασίζεται πρωτίστως στο αποτέλεσμα το οποίο στο συμπέρασμα ότι το Συμβούλιο ε, δεν πρέπει να βασίζεται σε μη ουσιώδη στοιχεία της συνθήκης του Σέγγεν και καταλήγει ότι από μια τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της συμφωνίας για το Σέγγεν θα πρέπει να θεσπιστούν νέα στοιχεία όσον αφορά το οργανισμό για τη Frontex. Τέλος, η σύσταση ε, οδηγεί σε μια διατήρηση του κανονισμού έως ότου υπάρξει ένα νέο νομοθέτημα σύμφωνα με τις ε, νομικές ε, διαδικασίες. Ε, όπως σας είπα, χαίρομαι που πραγματικά με τον τρόπο αυτό υποστηρίζεται η θέση την οποία εγώ υποστήριξα και η οποία εκφράζει και την άποψη της πολιτικής μου ομάδας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Πρόεδρε, επιτρέψατε μου να ξεκινήσω συγχαίροντας ιδιαίτερο τι νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και θα ήθελα να υπενθυμίσω τους συναντέλφους στην Επιτροπή αυτή ότι το Φεβρουάριο του 2010 ο κύριος Λόπεθ Αργγιλάρ απευθύνθηκε στις νομικές υπηρεσίες για νομική συμβουλή σε σχέση με αυτή την απόφαση του Συμβουλίου. Και στην περίπτωση αυτή η νομική υπηρεσία απάντησε το Μάρτιο του 2010 για να μας πει ότι στην περίπτωση αυτή η Επιτροπή ε, υπερεύει τις αρμοδιότητες της και άρα είναι δικαιολογημένη η προσφυγή στο δικαστήριο. Ε, συνεπώς η Επιτροπή αυτή ε, προσπάθησε να προσβάλλει την απόφαση του δικαστηρίου και να το φέρει στην Ολομέλεια. Και για να το κάνουμε ζητήσαμε μια απόλυτη πλειοψηφία στην Ολομέλεια. Και ε, το ψήφισμα υποστηρίχθηκε από 339 ψήφους. Δηλαδή υπήρχαν 30 ψήφοι λιγότεροι για να πετύχουμε την απόλυτη πλειοψηφία. Και ε, το ψήφισμα στηρίχθηκε ε, με μεγάλη πλειοψηφία, αλλά όχι με απόλυτη πλειοψηφία και αυτό το λόγο η απόφαση του Συμβουλίου ε, δεν ήταν δυνατόν πολιτικά να απορριφθεί από το Κοινοβούλιο. Όπως είπε ο κ. Κάσμαν, κατά συνέπεια ε, ξαναερχόμαστε σε αυτή την Επιτροπή και ζητούμε να δούμε κατά πόσο θα έπρεπε ο κανονισμός αυτός να ε, επανεξεταστεί με το σκεπτικό ότι πραγματικά η, ε, η Κομισιόν υπερεύει τις αρμοδιότητές της. Δεν ε, συμφωνώ πολύ με τον τρόπο που διατύπωσε ο κύριος Κάσμα το ιστορικό, αλλά το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε σήμερα είναι ότι ο Γενικός Εισαγγελέας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αποδέχτηκε την συμβουλή που ε, το απίφθηναν οι δικές μας νομικές υπηρεσίες και με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να τη συγχαρώ και επίσης υποστήριξε τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και πράττοντας αυτό προτείνει ε, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ο κανονισμός αυτός να θεωρηθεί άκυρος. Όπως ξέρουμε όλοι, ο Γενικός ε, Εισαγγελέας ε, δεν μπορεί να πάρει από μόνο του μια απόφαση, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε την ε, τελική κρίση. Αλλά τώρα ε, περιχόμαστε στην εξή κατάσταση. Τι θα κάνουμε από εδώ και εξή. Είμαι κάπω απογοητευμένο που η Επιτροπή δεν ήθελε καν να παρέμβει σήμερα. Εγώ θα ανέμενα την Επιτροπή να μα αποκαλύψει τα σχέδιά τη υπό το πρίσμα αυτή τη ε, γνώμοδότηση του Γενικού Εισαγγελέα και εάν ε, δεν, ε, και εφόσον δεν συνέβη αυτό σήμερα, τότε θα πρέπει να συμβεί εφόσον αποφανθεί οριστικά ο Γενικός Εισαγγελέας γιατί ε, ο κανονισμός έχει θεωρηθεί άκυρος, αλλά σύμφωνα με το δικαστήριο ε, εξακολουθεί να ισχύει έως ότου τροποποιηθεί, έως ότου αλλάξει. Και ε, αυτή τη στιγμή αλλάξει, θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει το πλήρες δικαίωμα συναπόφασης. Και ακριβώς αυτή είναι η ουσία του θέματος, γιατί έχουμε κάποιους κανόνες που ακυρώνει το Συμβούλιο βάσει μιας εσφαλμένης ε, διαδικασίας η οποία ε, μας αφαιρεί πλήρως το δικαίωμα συναπόφασης που θα είχαμε για την τροποποίηση αυτών των κανόνων. Και αυτή είναι η ουσία του θέματος. Θα έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία και να τροποποιήσει αυτούς τους κανόνες, ούτως ώστε να τους κάνει πιο δίκαιος από ό,τι είναι σήμερα. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο τρόπος, ε, η κατεύθυνση όπου θα πρέπει να κινηθούμε και αυτή είναι η κάθαρη γραμμή που παίρνει ο Γενικός Εισαγγελέας και αυτή τη στιγμή σε κρυφή οριστικά υπόθεση ε, θα πρέπει η Επιτροπή να επανέλθει σε μας και να ε, αναθεωρήσει αυτούς τους κανόνες αποδίδοντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πλήρη αρμοδιότητα συναπόφασης ούτω ώστε να μπορέσει να καταθέσει τροπολογίες για να αλλάξει αυτούς τους ε, κανόνες και να μην περιορίζεται σε, σε μια απλή δυνατότητα να πει ναι ή όχι. Ε, θα ήθελα κλείνοντας να ευχαριστήσω και πάλι την νομική υπηρεσία για το εξαίρετο έργο της. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπουζούτιλ. Βλέπετε ότι όταν θα πρέπει να ζητάμε πιο συχνά τη γνωμοδότηση της ε, νομικής υπηρεσίας, γιατί κάνουν πολλά πράγματα. κύριος ε, Κόσμαν. Πρέπει να είμαστε πολύ σαφείς, γι' αυτό λοιπόν θα πω το εξή. Δεν ήταν ε, σωστή η αριθμή που έδωσε ο κύριος Μπουζούτιλ. 336 ψήφοι υπέρ, 253 κατά και 13 αποχές. Επομένως το 33 ε, ψήφι και όχι 30. Εν πάση περιπτώσει, περιμένω ότι η Επιτροπή θα είναι σε θέση να απαντήσει όταν θα έχει το δικαστήριο ε, ε, φτάσει στην τελική του ετοιμιγορία. Και επίσης για τα πρακτικά, ο Γενικός Εισαγγελέας ε, ασχολήθηκε με τη διαδικασία και για το, με το κατά πόσον εφαρμόστηκε η σωστή διαδικασία και ε, εκεί εστιάζεται η ετοιμιγωρία του, κυρίως στην διαδικασία. Όμως, καλωσορίζω αυτήν την ετοιμιγωρία, αυτή την απόφαση και χαίρομαι ιδιαίτερος που οι συστάσεις ε, λένε ότι θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν ε, να ισχύει ο θαλάσσιος νόμος των ε, θαλασσίων συνόρων δηλαδή. Θα πρέπει να φύγω και δεν με συγχωρήσετε. Δεν έχω ζητήσει, δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο. Επομένως μπορούμε να θεωρήσουμε ότι ολοκληρώνεται η συζήτηση Είμαστε λίγο πιο πριν από την ώρα μας, τελειώσαμε πιο γρήγορα.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 ε, βλέπω ότι είναι εγγεγραμμένα τα υπόλοιπα σημεία και κλεισμένο των θυρών και ζητώ να μάθω ποιος ε, ε, μετά από αίτημα τίνος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ θεωρώ και θέλω να καταγραφεί ότι φρονώ πως δεν υπήρχε λόγος να είναι και κλεισμένο των θυρών, είναι ανώφελο, αλλά εν πάση περιπτώσει αφού έχει γίνει αποδεκτό δεν μπορώ να πω τίποτα.